Περνάμε στην έκθεση Hannibal, σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός του στην ισότητα των φίλων. Η συγκίτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους και ιδίω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τις ομάδες και τις ΜΚΟ που έχουμε συνεργαστεί μαζί μας και όλα τα δίκτυα των ε, ενώσεων που αγωνίζονται κατά της πορνείας και της ελαθρεμπορίας ατόμων. Βασίζομαι σε δύο οδηγίες. Την οδηγία για τα θύματα βίας του 2012 και την οδηγία για τη λαθρεμπορία ατόμων το 2011. Είναι σαφές ότι η λαθρεμπορία οδηγεί στην πορνεία και η πορνεία βασίζεται στην λαθρεμπορία. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι ένα διαμεθοριακό θέμα και ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και υγειονομικές επιπτώσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χαίρομαι λοιπόν που έχω αυτή την ευκαιρία να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα αυτό. Υπήρξε ένα δύσκολο και αφιλεγόμενο θέμα. Γιατί η νομοθεσία σε σχέση με την πορνεία, σε σχέση με την γενική λαθρεμπορία ατόμων, και η στρατηγική μας για αυτά τα διαμεθοριακά θέματα είναι φυσικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και σωστό είναι αυτό. Αλλά τα συντάγματα και η νομοθεσία των κρατών μελών έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν κολλάζεται η πορνεία. Ενώ η ε, προτροπή σε πορνεία ή η λειτουργία οίκων ανοχής είναι ποινικά αδικήματα σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία η πορνεία είναι απόλυτα νόμιμη. Είναι λοιπόν δύσκολο το να έχουμε μια γενική ρύθμιση και η έκθεσή μας θα πρέπει να λάβει υπόψη την πολυμορφία εθνικών ε, παραδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα όμως είναι σαφές. Δηλαδή πολύ λίγες γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον κλάδο της πορνείας το κάνουν εθελοντικά, εκούσια. Όσο εργαζόμουν για αυτή την έκθεση, μίλησα με πολλές γυναίκες που εργάζονται στον τομέα αυτό και πολλές ενώσεις γυναικών. Δεν βρήκα ούτε μία γυναίκα η οποία διάλεξε ως επαγγελματικό κλάδο την πορνεία με ελεύθερο τρόπο. Πολλές από αυτές τις γυναίκες ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι 62% των γυναικών που είναι αντικείμενα λαθρεμπορίας είναι γυναίκες οι οποίες τη χάνουν εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολλές φορές νέες γυναίκες και κορίτσια ακόμα. Αυτό και μόνο του είναι αρκετά αποτρόπαιο. Πέραν της ε, περίπτωσης αυτής υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες είναι τοξικομανείς και υπάρχουν και πολλές ε, γυναίκες και εδώ είναι δύσκολες στατιστικές πολλές από τις γυναίκες που βρίσκονται στην πορνεία έχουν περάσει πολύ δύσκολη και ταραγμένη παιδική ηλικία και έχουν υποστεί κακοποίησης. Σε μια εποχή κρίσης πολλές γυναίκες στρέφονται κατά ανάγκη στην πορνεία για να αντιμετωπίσουν την ε, ένδια. Η πορνεία λοιπόν δεν είναι επιλογή, δεν είναι μια εργασία όπως οποιαδήποτε άλλη. Είναι μια δραστηριότητα που στρέφεται κατά της ισότητας των φύλων. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, να λάβουμε υπόψη το σκανδιναμικό μοντέλο όπου είναι ο αγοραστής σεξουαλικών υπηρεσιών ο οποίος πρέπει να κολλαστεί και όχι η προσφέρουσα σεξουαλικές υπηρεσίες. Αυτό έχει οδηγήσει από το 1999 μέχρι τώρα σε σημαντική μείωση κατά 50% του συνολικού όγκου της πορνείας πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πορνεία, την μειώνουμε. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να μειώσουμε την πορνεία είναι να μειώσουμε την ζήτηση για πορνεία και το καλύτερο υπόδειγμα για κάτι τέτοιο είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται στη Σουηδία. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση σε όλους σας να υποστηρίξετε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάνιμπαλ. Ερχόμαστε στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία και εδώ έχω περισσότερες από ό,τι συνήθως αιτήσει και δεν μπορώ να τις ικανοποιήσω όλες. Λαμβάνει υπόψη ποιοι έχουν λάβει υπόψη, έχουν λάβει το λόγο ήδη και λαμβάνει υπόψη και την εθνική ισορροπία. Δεν είναι το λόγο στην κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην προσπάθεια της συναδέλφου Χόνιμπαλ Ο όρος πορνεία πράγματι περιλαμβάνει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αγοράζει κανείς υπηρεσίες για την προσωπική του ευχαρίστηση είτε είναι νόμιμη η πορνεία, είτε είναι παράνομη, δεν αλλάζει κάτι. Το ανθρώπινο όν αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα. Ξέρω ότι έχω γνώμες ε, οι οποίες διαφωνούν με τις γνώμες συναδέλφων από χώρες όπου έχει νομιμοποιηθεί η δραστηριότητα αυτή και υπάρχουν και κοινωνικές ρυθμίσεις, ε, κοινοτικές ρυθμίσεις που αναγνωρίζουν την δραστηριότητα της πορνείας. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστούμε την κυρία Ζαμπόσκα. Κυρία Εστρέλα τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πορνεία αυτή τη στιγμή αφορά 40 με 45 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, στην μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, καρπός της ανισότητας των δύο φύλων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά γεννάνε την πορνεία. Και φυσικά η δραστηριότητα συνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα, με το τράφικινγκ και τη σώματεμπορία. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν με το φαινόμενο αυτό οι χώρες μέλη. Κάποιες χώρες θεωρούν ότι είναι μια απλή παραβίαση των γυναικείων δικαιωμάτων, άλλοι ομιλούν για σεξουαλική εκμετάλλευση, άλλες ότι οι γυναίκες πρέπει να αποφασίζουν για το τι θα κάνουν με το σώμα τους. Το σκανδιναβικό πρότυπο νομίζω είναι αυτό που είναι πιο κοντά στην αξιοπρέπεια της γυναίκας. Η πορνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι επάγγελμα. Συγγνώμη Νικό. Κυρία Λούνατσεκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Χάνιμπολ στην έκθεσή της κατά την άποψη της πλειοψηφίας της ομάδας μου παρουσιάζει μια μονομερή αντιμετώπιση και δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλήθη, την, ε, τον πολυπληθή τρόπο αντιμετώπισης που έχουμε, τον ποικίλο τρόπο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί άντρε πάρα πολύ συχνά βλέπουν τις γυναίκες σαν αντικείμενο και όχι ως ανθρώπινα όντα. Αλλά η ποινικοποίηση όπως στις κανένας χώρες δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ λαθρεμπορίας για σεξουαλική χρήση, ε, πορνείας και εργασία στο σεξουαλικό τομέα που προέρχεται από ατομική απόφαση. Ξέρω ότι κάποιες γυναίκες μπαίνουν στο σεξουαλικό αυτό τομέα λόγω της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν, αλλά είναι προσωπική τους επιλογή. Μαζί λοιπόν με μέλη άλλων πολιτικών ομάδων προτείνουμε ένα εναλλακτικό ψήφισμα το οποίο εστιάζει στην ευθύνη των κρατών μελών και στο να υπάρχουν στρατηγικέ εξόδου για τι γυναίκε οι οποίε θέλουν να φύγουν από την πορνεία. Παρακαλώ υποστηρίξτε αυτό το εναλλακτικό ψήφισμα. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Η κυρία Ζουμπέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 93% των ατόμων που εκπορνεύονται είναι οι Η πορνεία οδηγεί σε μια διαιώνιση τη ανισότητα ανδρών και γυναικών και είναι μια, μορφή βίαιη μεταχείριση. Είναι ένα παλιό επάγγελμα και μια παλιά μορφή βίας κατά των γυναικών που είναι αποτέλεσμα του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός θεωρεί ότι όλα είναι εμπορεύσιμα και αυτό περιλαμβάνει και την ε, στενή προσωπική σχέση. Αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν να είναι αντικείμενα. Στις χώρες όπου η πορνεία είναι ε, νόμιμη, γίνονται οι γυναίκες ουσιαστικά επιχειρηματίες της νύχτας. Όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν παραγωγικά για τη χώρα. Μια γυναίκα η οποία πουλά την αξιοπρέπειά της και το σώμα της σε ένα άνδρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εισφάλει απόλυτα. Μια τέτοια εμπορευματική αντιμετώπιση θα πρέπει ε, ποινικοποιεί τον αγοραστή και δεν κάνει τίποτα για να εξασφαλίσει την προστασία των γυναικών αυτών. Ευχαριστώ κύριε Σούπερ. Σιόμπρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της πορνείας, και σε αυτούς που την εκμεταλλεύονται, απαιτείται να υπάρχουν αυστηρές νομικές ρυθμίσεις που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Να ενθυμούμεθα επίσης ότι σε ορισμένους χώρους, σε ορισμένες χώρες συγγνώμη, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή. Αντίθετα όμως με την εφαρμογή της. Οι νομικές ρυθμίσεις Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται. Στην Πολωνία, στην χώρα μου, υπάρχει πορνεία, ιδιαίτερα προσφέρονται υπηρεσίες τέτοιου είδους στους οδηγούς των φορτηγών που περνούν από τις μεγάλους οδικούς άξονες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα τέτοιο απαράδεκτο φαινόμενο. Ευχαριστούμε η κυρία Μολμπάη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει τόνους εγγράφων για την εμπορία όντων και παράλληλα βλέπουμε ότι οι διοκτικές αρχές δείχνουν αδιαφορία έναντι των γυναικών. Στη Βουδαπέστη ο Διευθυντής της Αστυνομίας αρνήθηκε να οργανώσει ένα εκπαιδευτικό τμήμα για τους ε, αστυνομικούς και αξιωματικούς σχετικά με το θέμα αυτό. Και η αστυνομία στην Αυστρία δημιούργησε μια μεγάλη φασαρία διότι ε, φεύγουν από την Ουγγαρία προς την Αυστρία νέες γυναίκες και εξαφανίζονται και μήνες αργότερα αρνείται η αστυνομία να ε, διατάξει μια έρευνα παρότι υπάρχει υποψία βίας κατά των γυναικών και υποψία σωματεμπορίας. Γνωρίζετε τις πρακτικές αυτές και τι προτίθεστε να κάνετε. Ευχαριστώ τη συνάδελφα Μολβάη. Συνάδελφος Μπορείς. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji i sutenerstwa Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πορνεία είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα. Καλύτερη νομοθεσία θα μπορούσε να ε, βοηθήσει ώστε να επιβληθεί η νομοθεσία και να εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης χρειαζόμαστε και κάποιες στρατηγικές για τις γυναίκες που θέλουν να αποσυρθούν από την πορνεία. Σίγουρα η πορνεία σχετίζεται με τη φτώχεια και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή για να διασφαλίσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα που έχει διασυνοριακό χαρακτήρα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2011 στην Ευρώπη αποκτήσαμε νέα νομοθεσία για τα θέματα εμπορίας ανθρώπων. Και θεωρούμε ότι Πρόκειται περί εγκληματικής δραστηριότητας ε, όταν μιλάμε για την εμπορία ανθρώπων. Ε, το 2016 θα πρέπει να ε, υποβληθεί μια έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων και θα είναι πολύ χρήσιμο να γίνει μια σχετική έρευνα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το θέμα της ζήτησης για απορνία. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Χίτ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατ' και δίνουμε το λόγο στην Επίτροπο κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με ευχαριστίες στην κυρία Μέρι Χάνιμπαλ για την έκθεση πρωτοβουλίας της. Είναι φρικτές οι συνέπειες της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και λαθεμπορίας. Υπάρχουν πολλές ιστορίες παραπλάνησης νέων κοριτσιών και γυναικών που οδηγούνται στο να πουλάνε το σώμα τους, να κακοποιούνται, να δέρονται, πολλές φορές να έχουν πολιθήκη από τις οικογένειές τους. Θέλω να τονίσω σαφές ότι για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η λαθρεμπορία ανθρώπων είναι απαράδεκτη με κάθε τρόπο. Είναι μια χονδροειδής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Μας λένε πολλές φορές ότι είναι ένα κρυμμένο έγκλημα η λαθρεμπορία ανθρώπων. Αλλά το βλέπουμε με τα μάτια μας. Είναι κάτι που γίνεται κάτω από τη μύτη μας. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε είναι αυτοί που κινούν τα νήματα πίσω από το προσκήνιο, οι εγκληματίες που ελέγχουν αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Βλέπουμε λοιπόν και τη σχέση μεταξύ φύλου και λαθρεμπορίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, 96% των ε, θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι γυναίκες και κορίτσια. Και αυτό είναι μια τραγωδία για κάθε μια από αυτέ τι γυναίκε και τα κορίτσια. Και αυτό συνδέεται με τη συζήτηση που είχαμε για το προηγούμενο θέμα στην έκθεση της κυρίας Παρβάνοβα. Αναγνωρίζουμε επίσης το ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια καταλήγουν στην αγορά πορνείας όχι με θελοντική επιλογή υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της αγοράς της πορνείας. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι αδιαφυσβήτητοι και έχουν γίνει όλο και πιο σαφείς. Επίσης η Europol μας πληροφορεί τα περισσότερα θύματα σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης έχουν πάει, έχουν πάει με λαθρεμπορία σε χώρες όπου είναι ελεύθερη ή ρυθμιζόμενη η πορνεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει και μία φιλόδοξη οδηγία για τη λαθρεμπορία ατόμων και μια στατηγική συνοδευτικού χαρακτήρα για να αντιμετωπίσουμε τη διάσταση του φύλου και την ανάγκη να μειώσουμε την, τη ζήτηση ε, για λαθρεμπορία ατόμων. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η πρόληψη είναι ο κύριος πυλώνας αυτής της στρατηγικής γιατί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να μειώσουμε την ε, ζήτηση για σεξουαλική εκμεταλλεύση για να εκμεταλλευτούμε ένα μικρό κορίτσι ή να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει πορνογραφικό υλικό, αυτό γίνεται μονάχα αν υπάρχει ένας δυνητικός χρήστης ή αγοραστής ε, υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μειώσουμε και εν καιρό να εξαλείψουμε αυτή τη ζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γεώργιεβα. Κλείνει η συζήτηση και για το θέμα αυτό. Αύριο στις 12 θα γίνει ψηφοφορία. Τελευταίο θέμα της μέσης διάταξης για απόψε η έκθεση ΣΑΙΕ ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Εκτελεστική Επιτροπή. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος ΣΑΙΕΡ.